Καλώς ήρθατε λοιπόν. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση της 30 Μαΐου του 2012 επιβεβαίωσε τις εντολές ε, των βουλευτών από 18-2012, την κυρία Μινοδόρα Κλειδέτη και τον κύριο Άλτα Σούσα από 9 Μαΐου του 2012. Παρακαλώ λοιπόν να συμφωνήσουμε για την έγκριση των εντολών αυτών. Υπάρχει αντίρρηση. Επικυρώνουμε λοιπόν τις έντολες αυτές. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η ομάδα των Ελευθεριών και Δημοκρατών ε, έχουν